να προβούν σε ανακοίνωση. Για τρίτη εβδομάδα συνεχίζεται η αντίδραση των διευμηνέων στα νέα μέτρα τα οποία έλαβε μονομερός η διοίκηση εις βάρος τους και μέσα σε όλα έχουμε και την επιστράτευση πάρα πολλών συναδέλφων, κάτι το οποίο στοιχειοθετεί περιορισμό του δικαιώματος απεργίας φυσικά. Thank you. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Από τη δική μου πλευρά έχω και εγώ ανακοινώσεις και αλλαγές στην ημερήσια διάταξη, διότι το υπαριθμόν 10 θέμα, η ψηφοφορία, προτείνεται, ε, συγγνώμη, αναβάλλεται για αύριο στις 10 και 30 μετά από το υπαριθμόν 27 που είναι η ακρόαση. Το 15 θα συζητηθεί μετά από το 18. Θα συνεχίσουμε τώρα με το θέμα 17. Ακρόαση υποψηφίων για την θέση του εκτελεστικού διευθυντή του οργανισμού IPO. Ως γνωρίζετε, ο εκτελεστικός διευθυντής του γραφείου διορίζεται από το Συμβούλιο, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού EUIPO. Εδώ θα προσθέσω ωστόσο στο 17 και το ζήτημα 16 της ημερής διάταξης που λησμόνησα να αναφέρω χθε. Συμμετείχα στη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου και το περιεχόμενο των συζητήσεων του οποίου είχε δύο σκέλη, αφενός την προεπιλογή υποψηφιωτήτων και το αποτέλεσμα της προεπιλογής είναι οι δύο υποψηφιότητες που είναι παρούσες σήμερα εδώ παροιμήν. Το δεύτερο θέμα στην ημερήσια διάταξη στην συνάντηση αυτή στην Ισπανική Αλικάντε ήταν η ετήσια έκθεση του 2017 που ωστόσο τελικώς οδήγησε σε μια σειραφή επένων. για τον Αντώνιο Καμπίνος, ο οποίος ε, ολοκληρώνει εδώ τη σταδιοδρομία του. Και περί αυτού επρόκειτο εν τέλει σε αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου. Οφείλω να τονίσω ότι η έπαινη ήταν ομόφωνη. Ούτε μία φωνή δεν ακούστηκε αντίθετη με τους επένους για το έργο του Αντώνιο Καμπίνος. Όλοι λοιπόν φάνηκαν πολύ ικανοποιημένοι από την εργασία του προσώπου αυτού, ο οποίος με την εργασία του έχει βάλει υψηλά τον πύχη για τον διαδοχό του ανεξαρτήτως του ποια από τις υποψηφιότητες θα επικρατήσει σήμερα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στις 5 Ιουνίου κατέληξε σε κατάλογο δύο υποψηφίων, τον κύριο Κριστιαν και την κυρία Κάι Χέρμαντ που βρίσκονται παρόντες, ε, παρόντα τα πρόσωπα αυτά εδώ. Πριν το Συμβούλιο προχωρήσει στον διορισμό του νέου εκτελεστικού διευθυντή, το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει τα δύο πρόσωπα αυτά να προβούν σε δηλώσεις και να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Ε, θα ακούσουμε τους δύο επιλεχθέντες υποψηφίους, αρχίζοντας με ονομαστική σειρά, πρώτα τον κύριο Ασαμπό. Έχετε 10 λεπτά, κύριε, για την ε, παρουσίαση που επιθυμείτε να κάνετε. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή μου η πρόσκλησή σας για την υποψηφιότητά μου ως Γενικού Διευθυντή της ε, Υπηρεσίας Διπλωμάτων Τεχνίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το IPO. Ήδη είμαι εκεί από το 2011 και ελπίζω και είμαι υπερήφανος για την προσφορά μου. Η υποψηφιότητά μου αποτελεί τη συνέχεια του τρέχοντος στρατηγικού σχεδίου. Έχουν υπάρξει συνεχείς βελτιώσεις στη λειτουργία του IPO και θα πρέπει να διατηρηθεί η πορεία αυτή και στο μέλλον λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζούμε μία περίοδο οικονομικών εξελίξεων και πολιτικών αλλαγών, γεωπολιτικών αλλαγών και τις είδαμε στην τελευταία συνάντηση της ομάδας των 7 και των προβλημάτων ανάμεσα στα κράτη-μέλη όπως το θέμα του Brexit και οι αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό οι προκλήσεις λοιπόν για το IPO είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία στα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων να περάσει στο επόμενο επίπεδο, να ανταμετωπίσουμε την αύξηση των ετοιμάτων για τέτοιου είδους διπλώματα και κατοχυρώσεις και από τρίτες χώρες και θα πρέπει επίσης τα δικαιώματα αυτά να γίνονται σεβαστά και στην Ένωση και εκτός η πρώτη προτεραιότητα, η πορεία μετατροπής και σύγκλησης και ολοκλήρωσης του συστήματος χορήγησης ε, διπλωμάτων ε, προχωρά. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε επενδύσει περίπου 100 ε, εκατομμύρια στον τομέα της βελτίωσης των δυνατοτήτων μας. Η ποιότητα και η προβλεψιμότητα των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουμε προς τις επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων και τις μικρομεσαίες ελπίζω να μπορούν να βοηθούν πέρα από την εθνική καταγραφή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις δυνατότητες των επιχειρήσεων αυτών. Βελτιώνονται οι δυνατότητες και οι έρευνες την οποία έχουμε κάνει μέσω του παρατηρητηρίου μόνο το 9% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το IPO για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους. Θέλουμε το ποσοστό αυτό να αυξηθεί και εμπορικά και γενικότερα. Να βελτιώσουμε επίσης τις δυνατότητες επένδυσης σε περιπτώσεις μεταφοράς τεχνολογίας και δοκιμασίας νέων προϊόντων, όπως επίσης και ε, πολλαπλασιασμό των τοπικών και περιφερειακών γραφείων που είναι σε άμεση επαφή με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν τεχνητά εμπόδια στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να καλύψει το σύνολο του κύκλου έτσι ώστε να ευνοούμε, θα έλεγα, το κοινό καλό, να δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης και να αυξάνουμε τις εξαγωγές. Και θα πρέπει επίσης να ενισχύουμε και να εμπνέουμε και τις τοπικές υπηρεσίες, τις εθνικές υπηρεσίες, και να συνεργαζόμαστε και με όλα τα help desk της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας ε, και μιας και οι νέες εξελίξεις στην τεχνολογία είναι ουσιαστικά καθημερινές ε, θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε ακόμα περισσότερο. Η στρατηγική μας τα τελευταία 7 χρόνια μας έχει βοηθήσει να καλύψουμε την αύξηση κατά 35% σε 7 χρόνια των αιτήσεων για χορήγηση αδειών. Και αυτά γίνονται στα πλαίσια και της διοργανικής συμφωνίας. Έχουμε επίσης βελτιώσει το ψηφιακό περιβάλλον της, του IPO και έχουμε ακολουθήσει μια πολιτική διαχείριση ανθρωπίνων πόρων μέσω της αναγνώρισης της εμπειρογνωμοσύνης και των ικανοτήτων του προσωπικού. Ε, και από 10% γυναικών σε διευθυντικές θέσεις φτάσαμε το 37% σήμερα και ελπίζω στο τέλος της περίοδου μου να φτάσουμε το 50%. Ο έλεγχος των τεχνολογιών είναι κάτι το οποίο μας επέτρεψε να εξοικονομήσουμε και αρκετές δαπάνες. Ξέρουμε όμως ότι έρχονται και νέες δαπάνες και νέες αλλαγές, συγγνώμη, και υπάρχουν δυνατότητες ε, έτσι ώστε να καταστούμε πιο χρήσιμοι και πιο φιλικοί στους χρήστες. Πάρα πολλέ απλές δράσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται με αυτόματο τρόπο, αυτοματοποιημένο μάλλον τρόπο, και ελπίζω ότι οι βελτιώσεις θα γίνουν σαφείς τα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επανειδρυθούμε ουσιαστικά για να καλύψουμε τις ανάγκες της νέας εποχής που έρχεται γρήγορα. Το IPO θα πρέπει να αναλαμβάνει την προσπάθεια αναγνώρισης των θεμάτων γύρω από την πνευματική ιδιοκτησία. Ήδη έχουμε κάποια δίκτυα χορήγησης πιστοποίησης ιδιαίτερα και για τις νομικές υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου. Τα έχουμε συζητήσει αυτά για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για τις ε, ονομασίες τοπικής προέλευσης, ιδιαίτερα στον γεωργικό τομέα. Είμαστε μια τεχνική υπηρεσία προς όφελος ε, των χρηστών των συστημάτων πληροφορικής και εφόσον το θέλει η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο μπορούμε επίσης να κάνουμε ακόμα περαιτέρω βήματα για να βελτιώσουμε το, ε, τις δυνατότητες των συστημάτων καταγραφής. Πρέπει να ελέγξουμε λοιπόν τις νέες τεχνολογίες που καθίστανται ε, διαθέσιμες στον τομέα της ε, τεχνητής νοημοσύνης, των blockchains και των καινοτομιών. Γι' αυτό ακριβώς το παρατηρητήριο προσπαθεί να δει τι δυνατότητες υπάρχουν σε σχέση με την χρήση των blockchain για να ελέγχουμε τις παραβιάσεις της πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάτι το οποίο θα μπορεί επίσης να καλύπτει και τις ανάγκες σε όλη τη χρονική περίοδο σε σχέση με, την, με τις νέες τεχνικές αλλαγές και επιστημονικές αλλαγές θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και με χώρες όπως η Κίνα που δημιουργούν νέες προκλήσεις, απειλές αλλά και ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό απαιτεί περαιτέρω προσπάθειες και για τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα και τα διαχειριζόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επίσης και σωστότερες και στενότερες σχέσεις με τις διεθνείς οργανώσεις που καλύπτουν το πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι απαραίτητο οι χώρες οι οποίες λειτουργούν σε παγκοσμιοποιημένη βάση να λειτουργούν σε ένα απεριβάλλον προβλέψιμο και διαφανές. Έρχομαι τώρα στο θέμα της επιβολής των αποφάσεων αυτών. Ξέρετε ότι το παρατηρητήριο έχει προχωρήσει στη διατύπωση εκθέσεων που είναι κεντρικές στον τομέα του σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων. Έχουμε αναπτύξει επίσης στενή σχέση και με τη Europol, στηρίζουμε το κέντρο ηλεκτρονικού εγκλήματος της Europol. Οι δραστηριότητές μας ε, φυσικά μας φέρνουν κοντά και στις δραστηριότητες των αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων ελέγχου ε, των σύνορων. Πολλά μένει να γίνουν ακόμα σαν παράδειγμα όταν ενημερώνουμε για τα δικαιώματα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στις ε, υπηρεσίες επιβολής τάξης, τις τελωνιακές υπηρεσίες και τις συνοριακές υπηρεσίες. Ιδιαίτερα τώρα που προχωρά σε μια γενικότερη ε, παγκοσμιοποιημένη και ολοκληρωμένη πολιτική. Ε, εφόσον με βάλετε στη θέση αυτή, με διορίσετε στη θέση αυτή, θα συνεχίσω την πορεία ολοκλήρωσης και σταθεροποίησης των τελευταίων χρόνων. Ε, η εμπλοκή των χρηστών και η συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα, σεβόμενοι τους διακριτούς ρόλους των εθνικών υπηρεσιών, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσφέρω είναι 30 χρόνια εμπειρίας, στον τομέα αυτό, μεταξύ των οποίων 15 σε υψηλές θέσεις. Επίσης ε, μπορώ να εγγυηθώ την διαφάνεια, τον έλεγχο, την ποιότητα και τις δυνατότητες ε, όπως και, τον, ε, και εξοικονομήσεις δαπανών. Νομίζω ότι μπορούμε να προσαρμόσουμε τη λειτουργία του γραφείου στις ανάγκες των χρηστών και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σόμπο. Έχουμε τώρα λίγο χρόνο να θέσουμε ερωτήσεις εφόσον επιθυμούν κάποια μέλη. Επιθυμείτε να θέσετε κάποια ερώτηση στον κύριο Σάμπο. Έχει καλώ Μπορούμε να θέσουμε ερωτήσεις και μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης παρουσιάσεως. Στην οποία περίπτωση, κυρία Χέρμαν, θα θέλατε να λάβετε τον λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμες κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, θα ήθελα να σας δείξω ότι στη φωτογραφία αυτό το ρομπότ που κάνει delivery γευμάτων, λουλουδιών, δεμάτων. Για την ώρα πάντως αυτό που κάνει είναι να κάνει delivery της παρουσίασής μου. Ελπίζω ότι η συσκευή θα λειτουργήσει και θα αλλάξει διαφάνεια, οπότε θα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Συνεχίζει η Χέρμαντ. Στην διαφάνεια αυτή ε, βλέπετε τις προκλήσεις και τις παγκόσμιες τάσεις όπως τις βλέπω εγώ. Η νέα οικονομία, οικονομία που βασίζεται στο sharing, στο να συμμετέχουν όλοι. Νέες μορφές εργασίας, όπως οι εικονικές συνεργασίες, δηλαδή οι πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν μαζί σε ε, δίκτυα και νέες γενιές που εργάζονται, νέες τεχνολογίες από τις οποίες μερικές γνωρίζουμε, άλλες μας είναι ακόμη άγνωστες, αλλά επινοούνται κάθε μέρα και νέες. Και εδώ βλέπετε εμένα στην διαφάνεια αυτή που δείχνω αυτή τη στιγμή. Είμαι πανεπιστημιακή, ε, είμαι πανεπιστημιακός δάσκαλος, είμαι ε, δικαστής και ταυτόχρονα ε, διέπομαι από πνεύμα καινοτομία και ε, λαμβάνω πολιτικές αποφάσεις. Είμαι μια πραγματική ηλεκτρονική εστονή, για να σας το πω έτσι, ε, που έχω εμπλακεί στην ανάπτυξη του συστήματός μας, στη χώρα μας δηλαδή, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όχι μόνο στο δικαστικό σώμα, αλλά και γενικότερα στο δημόσιο από το 2005. Έχω λοιπόν εμπειρία στον τομέα αυτό. Στην ετήσια κοινή διακήρυξη των νομοθετικών πρωτοβουλειών, τα τρία θεσμικά όργανα, Επιτροπή, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, συμφώνησαν σε έναν αριθμό θεμάτων που συνδέονται με το έργο του οργανισμού EU IPO, του Γραφείου Σημάτων δηλαδή. Ας αρχίσουμε με την προστασία της ασφάλειας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όλες και όλοι γνωρίζουμε ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις και οι διάφορες εγκληματικές ομάδες χρηματοδοτούνται εν μέρη από την πώληση ε, πλαστών προϊόντων. Έχουμε νέα όθηση σε επενδύσεις και ε, στην απασχόληση και ανάγκη από τέτοιες. 38% όλων των θέσεων απασχόλησης, πάνω από το 1 τρίτο δηλαδή, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σχέση με την ηλεκτρονική τεχνολογία. Έχουμε επίσης μπροστά μας την εφαρμογή της ψηφιακής ενίας αγοράς, την ψηφιοποίηση της παροχής υπηρεσιών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια και των θεσμικών της οργάνων. Παρόλο που μπορώ να πω ότι η ψηφιοποίηση ίσως να μην είναι χθεσινό πρόβλημα, είναι σημερινό πρόβλημα για αύριο, για το μέλλον, για το προσεχές μέλλον δηλαδή θα πρέπει να ε, προβληματιστούμε και να, ε, σκεφτούμε τις ε, αυτοματοποιημένες τεχνολογίες προσφοράς υπηρεσιών. Και το ίδιο απειό είναι ένας άξονας, ένας οργανισμός γύρω από τον οποίο στρέφονται πολλά από τα πράγματα αυτά και εταίρος των νομοθετικών οργάνων για να προσφέρει γνώση βασισμένη και θεμελιωμένη γερά σε ενδεικτικά και αποδεικτικά στοιχεία για την εξέλιξη των ηλεκτρονικών τεχνολογιών και της ε, διανοητικής ιδιοκτησίας και να προωθήσει διάφορα ε, project ε, συνεργασίας και άλλες δραστηριότητες. Νομίζω ότι ο οργανισμός EU IPO θα πρέπει να έχει την ικανότητα να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την εκπαίδευση και βεβαίως να αναλάβει και νέες ευθύνες συζητήσατε σήμερα το πρωί άλλωστε μια επιλογή μέσα στα πλαίσια της πρότασης για την οδηγία για το copyright να δημιουργηθεί ε, μια δημόσια δικτυακή πύλη για την πρόθεση της πολιτισμικής ποικιλομορφία. Για να, ε, για να υλοποιηθεί το όραμα αυτό, χρειαζόμαστε πρώτα-πρώτα τους κατάλληλους ανθρώπους σημαίνει ανθρώπους που θα είναι αφοσιωμένοι στο έργο τους γιατί οι άνθρωποι είναι και το, το ανθρώπινο δυναμικό είναι και ο μεγαλύτερος πλούτος οποιοδήποτε οργανισμού. Πρόκειται για μια πρόκληση να φέρει κανείς δηλαδή κοντά τις διάφορες γενναίες για να συνεργαστούν. Είναι πρόκληση να διασφαλίσει κανείς ότι και το τελευταίο μέλος του προσωπικού κάνει δουλειά που ε, να του φαίνεται ενδιαφέρουσα και ε, να ε, θεωρεί ότι αξίζει. Και επομένως είναι και η πρόκληση για το management να βρει την καλύτερη δυνατή θέση όπου μπορεί να αποδώσει το κάθε μέλος του προσωπικού. Και βέβαια χρειαζόμαστε μια οργάνωση δομημένη σε μια δομή που θα στηρίζει και θα προωθεί και την προσωπική πρωτοβουλία, αλλά και την διάθεση να επιτύχει κανείς συγκεκριμένους στόχους στην σταδιοδρομία του και να στηρίζει κάθε δημιουργική ιδέα. Όχι μόνο η δομή, αλλά και το στυλ της διοίκησης είναι σημαντικά. Δηλαδή χρειάζονται ξεκάθαρες ευθύνες και ξεκάθαροι πόροι που να επιτρέψουν τη λειτουργία του οργανισμού. Η διοίκηση του οργανισμού οφείλει να διασφαλίσει ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ξεκάθαρη και διαφανής ώστε να μπορεί να στηριχτεί πάνω σε αυτήν η ανάπτυξη. Και βεβαίως, ο οργανισμός EUIPO θα πρέπει να παίξει πρωτοπόρο ρόλο για την τεχνολογική ανάπτυξη. Όταν ακούμε ότι θα φτιάξουν αυτή την εβδομάδα ένα απλόκαθον, έναν αγώνα για την σύγκριση σχετικών τεχνολογιών. Στην Εστονία έχουμε χρησιμοποιήσει την τεχνολογία blockchain, θα είναι ένας μαραθώνιος blockchain δηλαδή, ήδη από το 2012. Άρα έχουμε έξι χρόνια ήδη εμπειρίας Νομίζω ότι είναι ο σωστός δρόμος πρέπει να ακολουθήσουμε, όμως από την άλλη μεριά υπάρχουν και πολλά πράγματα που μένουν να γίνουν ακόμη. Δεν βλέπω σχέδιο, για παράδειγμα, για ψηφιακή ταυτοποίηση. Παρόλο που έχουμε σχετικό κανονισμό που θα αρχίσει να ισχύει από τον επόμενο Ιανουάριο. Αυτή τη γνώση την διαθέτω και μπορώ να την φέρω στην εργασία μου αν αναλάβω την ε, θέση στο Αλικάντε και να βοηθήσω να ξεπεραστούν και οι στόχοι των προγραμμάτων που έχουμε ως τώρα. Όλα αυτά βέβαια δεν μπορούν να γίνουν χωρίς συνεργασία. Ακούσαμε ότι 9% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μόνο κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους διανοητικής ιδιοκτησίας. Πρόκειται λοιπόν για ένα τεράστιο τομέα που πρέπει να καλλιεργηθεί. Ε, σημαίνει αυτό συνεργασία μεταξύ βιομηχανιών, μεταξύ οργανώσεων βιομηχανιών. Ε, σημαίνει επίσης συνεργασία με πανεπιστήμια, με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πρόκειται για συνεργασία επίσης μεταξύ των εθνικών γραφείων ε, διανοητικής ιδιοκτησίας και του EU IPO, διότι γνωρίζετε στον κανονισμό για τα εμπορικά σήματα το ευρωπαϊκό σύστημα προβλέπει συνεργασία του EU IPO με τα εθνικά γραφεία ε, διανοητικής ή πνευματική και εφόσον αυτά αποτελούν μία ενότητα. Βεβαίως σημαίνει επίσης και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο Υπουργών. Και τέλος η σπουδαία ερώτηση του εκατομμυρίου δολαρίων. Τι θα κάνουμε με τα χρήματα. Εάν πάρουμε για παράδειγμα το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο στη νέα πρόταση που γίνεται, που δίνει έμφαση στην εκπαίδευση, στην καινοτομία και στην ανάπτυξη. Αν πάρουμε και τις νομοθετικές προτεραιότητες στην κοινή δήλωση των θεσμικών οργάνων και από την άλλη μεριά τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Γραφείου Σημάτων του Αλικάντη. Και αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, αυτά μας δίνουν την απάντηση στο ερώτημα που έκανα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου και πολύ ευχαρίστως είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Thank you very much. σας ευχαριστώ πολύ. Mr. Καβαντά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά ε, τους ε, δύο προλαλήσαντες. Θα ήθελα να καταλάβω εάν ε, είχατε το χρόνο να σκεφτείτε σοβαρά το θέμα της συνεργασίας με τα τελωνία, γιατί θεωρώ ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σπουδαίο σημείο και θέμα. Ε, στην Ευρώπη έχουμε αποτελεσματικό και τελωνιακές οργανώσεις, ας πούμε αυτή της, ε, τα τελωνία της Ισπανίας. Ε, υπάρχουν όμως και άλλα τελωνία τα, και υπηρεσίες όπως αυτή της Πολωνίας που δεν είναι στελεχωμένα με αρκετό προσωπικό και υποφέρουν. Ε, ξέρω ας πούμε ότι στην Ανατολική Πολωνία υπάρχει ε, ένα σταθμός όπου οι τελωνιακοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να βλέπουν τα κινέζικα τρένα να περνούν ή τα τρένα με τα κινέζικα προϊόντα. Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου φαίνεται ότι η ελληνική αστυνομία δεν έχει πλέον δικαίωμα να μπει στο λιμάνι του Πειραιά. Ε, υπάρχουν επομένως ε, κάποιες, ε, ε, ε, κάποιες περιοχές τις οποίες λιμένονται διάφοροι. Επομένως, ερώτηση. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι μπορείτε σε αυτό το νευραλγική σημασίας και ουσιώδου σημασίας θέμα ε, μπορείτε να προωθήσετε ε, τη συνεργασία με τα τελωνία. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε, ρωτά ο πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ, λέει η κυρία Χέρμαντ. Πιστεύω ότι εδώ έχουμε δύο διαστάσεις. Πρώτα απ' όλα, ακράδαντα πιστεύω ε, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αποτελεσματική εργασία σημαίνει ότι ε, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Επομένως, ναι, βεβαίως ε, η καλή εκτέλεση προϋποθέτει καλή εκπαίδευση. Εκπαιδεύεις, καταρτίζεις ανθρώπους που πρέπει να καταλάβουν, να γνωρίζουν πώς είναι οι διαδικασίες και ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους. Τι πρέπει να κάνουν ακριβώς. Υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο είναι δυσκολότερο και αφορά τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών και όχι μόνο. Πιστεύω ότι ο αγώνας, αν θέλετε, αυτή η μάχη κατά των παραποιημένων προϊόντων ξεκινάει από αμοιβαία αναγνώριση των προβλημάτων από Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, δεν πρέπει απλώς η υπηρεσία πνευματική, ο οργανισμός πνευματικής ε, διανοητικής διοκτησίας που θα πρέπει να αντιμετωπίσει μόνος του το πρόβλημα. Οι, οι χώρες μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. για οποιοδήποτε πρόβλημα. Εάν προκύψει πολιτική δέσμευση, τότε και η εκτέλεση θα είναι καλή. Ο κύριος Ασαμπό, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρόβλημα και η λύση του Ε, μάλλον για να λυθεί το πρόβλημα χρειάζεται ε, πολυμερής και πολυεπίπεδη προσέγγιση. Όπως είπε και η κυρία Χέρμαντ, ε, πρέπει να προκύψει πολιτική συμφωνία σε υψηλό επίπεδο έτσι ώστε να ε, συνεχίσει ο αγώνας ε, κατά των παραποιημένων προϊόντων και επίσης χωρίς πόρους κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί είναι χωρίς όπλα και τα κράτη-μέλη το αποφασίζουν αυτό το κατά πόσο δηλαδή δίνουν τις, τους πόρους. Βέβαια οι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο αποτελεσματικό και στοχευμένο είναι αδύνατον να ε, ε, ψάξει κανείς και να ελέγξει κάθε μικρό δέμα που περνάει τα σύνορα. Χρειάζεται συγκεκριμένη στοχευμένη έρευνα που σημαίνει ε, πληροφορίες, intelligence ε, και δυνατότητες ταυτοποίησης των προβληματικών δεμάτων. Όσον αφορά ε, τις πληροφορίες, όπως είπα και στην ε, εισήγησή μου έχουμε στοχευμένες δράσεις μαζί με την Europol ε, έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε στη ρίζα ε, το φαινόμενο της μεταφοράς παραποιημένων προϊόντων. Υπάρχουν, έχουμε επίσης δυνατότητες διαχωρισμού, ταυτοποίησης του αυθεντικού προϊόντος σε αντιπαράθεση με το ε, παραποιημένο και επίσης ε, ε, ζητούμε και έχουμε επαφές με τις εταιρείες παραγωγής που μας δίνουν κάποια στοιχεία και όλα τα οτιδήποτε γνωρίζουν όσον αφορά όσον αφορά τις διαδρομές που ακολουθούν τα ύποπτα πακέτα. Τώρα, επιτόπου Βεβαίως ε, χρειάζονται καταρτισμένοι ε, αξιωματικοί και καταρτισμένο προσωπικό γενικά. Στην Ακαδημία και στο Παρατηρητήριο έχουμε δημιουργήσει ε, εργαλεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους ε, υπαλλήλου ε, ε, για να αναγνωρίζουν ευκολότερα και αποτελεσματικότερα τα παραποιημένα προϊόντα. Επομένως καταλαβαίνετε ότι για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτά τα παραποιημένα προϊόντα, τα προϊόντα απομίμησης, χρειάζεται πολυεπίπεδη προσέγγιση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλετε συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Καβαντά, παρακαλώ. Κατάλαβα καλά Κύριε Σόμπο, αναφέρεστε στις επιχειρήσεις. Έχετε την πρόθεση να διευρύνετε τα μέσα καταπολέμησης των απατών όχι μόνο με τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πιστώσεις της Επιτροπής δηλαδή, αλλά και με ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία θέλουν να δώσουν οι επιχειρήσεις έτσι ώστε να ενισχυθεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας των αυθεντικών τους προϊόντων. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοώ όταν λέω συντονισμένη δράση. Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι, είτε οι αρχές enforcement λέει στα αγγλικά ο μιλητής, όπως και οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων που επιθυμούν να υπερασπιστούν τα προϊόντα τους από την παραποίηση ε, να συνεργαστούν. Αν δεν γίνει αυτό δεν θα το πετύχουμε. Μία ερώτηση επιπλέον λέει ο Η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νομίζω θα συμφωνήσουμε. Αν δείτε την κατάσταση σήμερα, πιστεύετε ότι τα βασικά προβλήματα βρίσκονται στον τομέα της εφαρμογής των ρυθμίσεων ή μήπω ότι να υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα κεφάλαιο, θα έλεγα, νομικό, το οποίο να ελείπει και πρέπει να καλυφθεί έτσι ώστε η Ευρώπη να σημειώσει ε, βήματα πρόοδου. Η ερώτηση απευθύνεται και στους δύο φυσικά. Σε επίπεδο νομοθετικό, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα ενιαίο, ε, ενιαίο σύστημα χορήγησης διπλωμάτων είναι κάτι το οποίο θα μειώσει το κόστος της καταχώρησης και προστασίας. Απαιτείται χρόνος όμως γι' αυτό. Σχετικά με τα υπόλοιπα δικαιώματα, νομίζω ότι οι προκλήσεις τις οποίες εντοπίσαμε ήδη, όπως η σύγχρονη τεχνολογία και η ισχύουσα νομοθεσία να καταστήσει βατή με τον 21ο αιώνα σε επίπεδο τεχνολογίας είναι και αυτό κάτι το πολύ σημαντικό. Σαν παράδειγμα ο κανονισμός για τη σχεδίαση προϊόντων που είναι υπό αναθεώρηση υπάρχει πάντα ένας κανονισμός εδώ ο οποίος δεν καλύπτει αυτά τα οποία συζητήσατε το πρωί όπως την τρισδιάστατη εκτύπωση. Δεν υπάρχουν ε, μειώσεις κόστους για την σόρευση δεδομένων ηλεκτρονικά. Ε, οι, οι βασικές ε, θα έλεγα νομοθεσίες ε, χρήζουν ενημέρωσης και επικαιροποίησης. Σας ευχαριστώ. Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν νομίζω ότι μας διαφεύγει κάτι όταν μιλάμε για ενιαίο σύστημα ευρεσιτεχνίας ή κατάθεση σχεδίων ευρεσιτεχνίας το θέμα είναι περισσότερο θέμα εφαρμογής των κανόνων που ισχύουν. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στο σύστημα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ δημοφιλές σαν ιδέα, αλλά στην Ευρώπη μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια και το πρόβλημα στην Ευρώπη είναι περισσότερο θέμα εφαρμογής. ισότιμης εφαρμογής, έτσι ώστε κάθε κράτος μέλος να εξετάζει τις ανάγκες τις οποίες έχει και κάθε κράτος μέλος να μην επαφίεται αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην εξαρτάται μόνο, ε, να μην βοηθά μόνο σε επίπεδο χρηματικό, αλλά και σε επίπεδο ανθρώπινο δυναμικό. Τίθεται λοιπόν το θέμα της εφαρμογής. Καλώς, ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που έχει ζητήσει το λόγο. Αυτό σημαίνει ότι θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την παρουσία σας εδώ. Αγαπητοί υποψήφοι, συνυποψήφοι, να σας ευχηθώ καλή τύχη σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, επαναλαμβάνω εδώ σήμερα. Για έναν από εσά προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά.